Ας ξεκινήσουμε. Λυπούμε για την ε, καθυστέρηση. Υπήρχαν προβλήματα οργανωτικά. Τέλο πάντων, θα ξεκινήσουμε έγκριση λοιπόν του σχεδίου της ημερήσιας διάταξης. Έχει διανεμηθεί αν δεν έχετε να προτείνετε κάτι, αν δεν έχετε αντιρρήσεις, αν δεν θέλετε κάτι να προσθεθεί, μπορεί να εγκριθεί όσο έχει τροποποιηθεί. Αυτή η συνεδρίαση μεταδίδεται στο διαδίκτυο μέσω web streaming. Καλωσορίζουμε λοιπόν ακροατές θεατές. Έχουμε και το newsletter IMCO που δημοσιεύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Αντίγραφα μπορείτε να τα βρείτε εκεί δίπλα στην είσοδο της αίθουσάς μας. Μπορείτε όμως να μπείτε και στο δίκτυο των φίλων του, της ΕΜΚΟ με το να γραφείτε συνδρομητές στο newsletter και να σας αποστέλλετε ηλεκτρονικά. Επόμενο σημείο είναι η έγκριση των πρακτικών. Θα συνεχίσουμε και θα πάμε στο 5, 27η της έκθεση για παρακολούθηση του, κατά πόσο, του πώς εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό δίκαιο. Θα δώσω το λόγο στον Κρίσιαν Μπουσόλ, τον εισηγητή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η δεύτερη εκθεση για παρακολουθηση του κατα ποσο το πως εφαρμοζεται το ευρωπαικο δικαιο θα δωσω το λογο στον κρισιαν μπουσολ τον εισηγητη ευχαριστω παρα πολυ κυρια προεδρε κυρια προεδρε αγαπητοι συναδελφοι ειναι η δευτερη της εκθεση για την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου και χαίρομαι που μου δίνεται δυνατότητα να κάνω σύγκριση της προόδου που επιτυγχάνεται από έτος σε έτος είναι κάτι που ήδη συζητήσαμε όταν υιοθετήσαμε την έκθεση της κυρίας Καλιέντε για τη διακυβέρνηση και την εταιρική συνεργασία στην ενιαία αγορά, μια σημαντική συζήτηση που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη επίση και για την σημερινή μα συζήτηση. Η σωστή εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου είναι κρισίμου σημασία, ώστε να εγγυηθούμε την εύρυθμη λειτουργία τη ενιαία αγορά. Εάν συγκρίνουμε το 2008 με το 2009, παρατηρούμε κάποια πρόοδο, αλλά για να είμαστε ειλικρινεί, τίποτα ιδιαίτερα θεματικό. Διαβάζοντα αυτή την έκθεση, μου δημιουργείται ένα συνέστημα του déjà ότι ήδη τα έχω δει αυτά. Είναι απογοητευτικό. Σε κάποιου τομεί χρειάζονται προσπάθειε, τα επαγγελματικά προσόντα, οι, οι υπηρεσίε, οι κρατικέ προμήθειε. Ε, είναι μερικοί τομεί που θέλουν βελτίωση. Είναι συνεχώ αναδυόμενα θέματα που σημαίνει ότι κάτι πρέπει να γίνει ούτω ώστε να ε, σημειωθεί πρόοδος στον τομέα αυτόν. Όμως ε, νομίζω ότι έχουμε λόγους ε, να είμαστε ακόμα αισιόδοξοι, διότι έχουν βελτιωθεί κάπως τα πράγματα. Φερρυπίν, ο μέσος όρος της, των υποθέσεων καθυστερημένης εσωμάτωσης στο Εθνικό Δίκαιο πήγε από 55% στο 51%. Πιο γενικά, οι διαδικασίες προς παράβαση χρειάζονται λιγότερο χρόνο από ό,τι στην περασμένη δεκαετία, αλλά ο αριθμός των υποθέσεων παραβάσεων είναι υψηλό, άρα μπορούν να επέλθουν περαιτέρω βελτιώσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει να διστάσει να χρησιμοποιεί τι δυνατότητε που εισάγει η συνθήκη τη Λισαβόνα, ούτω ώστε να ζητήσει επιβολή οικονομικών κυρώσεων από το πρώτο στάδιο, δεν υπάρχει καμία άλλη λύση, για να πείσει τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν το κοινοτικό δίκαιο με πιο σοβαρό τρόπο. Εξακολουθεί να χρειάζεται πολύ χρόνο για τι διαδικασίε κατά παράβαση και καλωσορίζει το δυνατόν ότι το πιλωτικό πρόγραμμα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, τα πιλωτικά προγράμματα του έλξαν περισσότερα κράτη-μέλη. Αυτό αφορά συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κράτη-μέλη. Και αυτό μπορεί να βοηθήσει την επίλυση των προβλημάτων σε ένα πρώιμο στάδιο και έτσι θα αποφευθούν οι παραβιάσει. Για να αποφευθεί η λανθασμένη εφαρμογή των ε, νόμων, μπορεί να κάνουν κάτι θεσμικά τη Ευρωπαϊκή Πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί όταν συντάσσουμε, θεσπίζουμε νομοθεσία και να προσπαθήσουμε να είμαστε σαφέστεροι και ακριβέστεροι. Αυτό θα αύξανε την ασφάλεια δικαίου και οι δημόσιες αρχές θα μπορούν να καταλαβαίνουν καλύτερα το κοινοτικό δίκαιο. Οι πίνακε συσχετισμών μπορούν να βοηθήσουν τα μάλα διότι παρέχουν μεγαλύτερη ευκρίνεια και επιτρέπουν τη σωστή παρακολούθηση τη εφαρμογή τη νομοθεσία περί αγορά. Μια άλλη ιδέα που καλωσορίζω είναι η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων που θα συμπεριλαμβάνει νομοθεσία και νομολογία για θέμητες εμπορικές πρακτικές. Τέτοια βάση δεδομένων μπορεί να είναι χρησιμότατη και για τις δημόσιες αρχές και για τους πολίτες και πιστεύω ότι η εφαρμογή αυτών ε, των μέτρων και σε άλλου τομεί είναι κάτι πολύ χρήσιμο. Και τα στοιχεία από του πίνακε συσχετισμού ε, θα μπορούν να ενταχθούν σε βάσει δεδομένων για την αύξηση ε, τη διαφάνεια. Και κάτι εξίσου σημαντικό στο τέλο, θα ήθελα να επαναλάβω την υποστήριξή μου για την περαιτέρω ανάπτυξη του Solvit και του Europe Portal ούτω ώστε μέσω αυτής της θύρας να μπορούν να έχουν πρόσβαση οι πολίτες και να λύσουν τα προβλήματά τους που προκύπτουν από έλλειψη εφαρμογής ή λανθασμένη εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη ε, τα όρια που τίθενται για το κείμενο, για το σχέδιο γνωμοδότησης, το κείμενό μου δεν είναι εξαντλητικό, θα μπορούσα να το βελτιώσω, θα μπορούσα να βελτιωθεί, γι' αυτό θα είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένο αν μου πείτε ποιε είναι οι απόψει σα και αν μου υποβάλλουν οι σκιώδει εισηγητέ διάφορε τροπολογίε ή και άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι θα έχουν σαν σκοπό τη βελτίωση τη γνωμοδοτήσεως. Αυτά λοιπόν και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε θα δώσουμε στους σκιώδεις εισηγητές ε, το λόγο στον κύριο Σουάμπ, εκπρόσωπος του ΕΛΚ. Μήπως θέλετε να εκφράσει την άποψη του ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ τον συνάδελφο κύριο Μπουζό για την διευκρίνηση ε, των δυσκολιών ε, που σημειώνονται στη μεταφορά στα εθνικά δίκαια. Επίσης, ε, το θέμα των ε, παραβιάσεων του κοινοτικού δικαίου είναι ένα συναφές ε, πρόβλημα, διότι άπτεται της χρονικής διάρκειας των διαδικασιών για να ξεκινήσει η διαδικασία προσφυγής μέχρι ότου ε, βγει τελική απόφαση ε, για το κοινοτικό δίκαιο αν υπάρχει παράβαση ή όχι λαβή υπερβολικός χρόνος και αυτό δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό και πρέπει να βελτιωθεί. Αυτά που προτείνει ο κ. Μπουζό είναι εύλογα και εφικτά και την υποστηρίζουμε την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία, η κυρία Μαρία Πέρες έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να ευχαριστήσω τον κύριο Μπουσό για την δουλειά του και το εξαιρετικό κείμενο που μας παρουσίασε σήμερα, το οποίο περιλαμβάνει τα σημαντικότερα σημεία, τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει η γνωμοδότησή μας. Και με τον επικοδηγωματική αυτή θέση, ε, θα ήθελα όμω να προσθέσω και κάποιε ιδέε εγώ. Πρώτον, πρέπει να επιμείνουμε στη σημασία του να ενδυναμώσουμε την συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών ε, θεσμών και των κρατών μελών, όπω ε, ανέφερε ο κ. Μπουσόη. Επιπλέον, θα πρέπει να προωθήσουμε, να ψάξουμε για εναλλακτικά μέσα που θα μας επιτρέψουν να, να, να, να βοηθήσουμε την εφαρμογή της νομοθεσίας με στόχο ε, να μην ε, ε, υπάρξει ένα κορεσμό στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Επιπλέον θα πρέπει να ενισχύσουμε τη, τα θέσμα, τα θεσμικά μέσα όπως το Solvit και το, και το Pilot. Επιπλέον θα πρέπει να απαντήσουμε σε μια παλιά σε κάτι που έχουν ζητήσει οι πολίτες από παλιά για την ε, επίλυση των συγκρούσεων. Τέλος, θα πρέπει να επιμείνουμε να υπάρξουν οι, οι πίνακες συσχετισμών για να μπορέσουν ε, να κάνουμε την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μποσό για την εξαιρετική του δουλειά και στην ομάδα μου θα παρουσιάσω ορισμένε τροπολογίε και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα. Ευχαριστώ κυρία Ρούλε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συντάκτη του σχεδίου έκθεσης για την εξαιρετική συνεργασία και για την ε, πάρα πολύ καλή έκθεση την οποία υποστηρίζω. Έχω ε, ορισμένες δευτερεύουσες παρατηρήσεις και μικρές αλλαγές που θα ήθελα να κάνω. Όπως είπε και ο εισηγητής υπάρχει και το πρόβλημα της έκτασης της έκθεσης αυτής εγώ θα ήθελα να τονίσω τη διαφάνεια για την υφιστάμενη κατάσταση της, ε, των διαδικασιών, διότι πολλές φορές γίνομαι ε, γνώστης παραπώνων ότι δεν ενημερώνονται έγκαιρα ε, τα αρμόδια πρόσωπα, τα αρμόδια στελέχη και οι αρχές από την Κομισιόν ότι υπάρχει το ε, α ή το β πρόβλημα. Θέλω λοιπόν απόλυτη διαφάνεια και στο σημείο 5 πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε μία μικρή προσθήκη και να πούμε ότι αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες της Εκτελεστικής Επιτροπής ιδιαίτερα στην αναγνώριση ε, επαγγελματικών ικανοτήτων και στην ε, ε, σύνταξη αποφάσεων με απόλυτη σαφήνεια και καθαρότητα. Ε, κάτι τέτοιο, δηλαδή. Να ευχαριστήσουμε την Εκτελεστική Επιτροπή. Μια μικρή προσθήκη και κατά τα άλλα υποστηρίζω την έκθεση και ευχαριστώ τον εισηγητή για τις προσπάθειες του. Θαυμάσια έκθεση. Ευχαριστώ. Έχω την εντύπωση, λέει η Πρόεδρος, ότι αυτό το θέμα δεν ξεσηκώνει έναν τεράστιο ενθουσιασμό ε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κανείς εδώ από το κόμμα των Ευρωπαίων Συντηρητικών όχι τότε από την ΓΚΟΕ ε, άλλος ε, εκπρόσωπος πολιτικής ομάδας όχι, ωραία υπεσημεί κάποιο άλλο μέλος της Επιτροπής μας να μιλήσει ο, εντάξει, ησυχία Καλύτερα... Α, η Επιτροπή. Η Επιτροπή θα έχει τίποτα να πει. Ο κύριος Κάρ. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ είμαι ε, παθιασμένος <laughs> για αυτήν την έκθεση διότι μετά από αίτηση το Κοινοβουλίο έγινε αυτή η έκθεση και μας δίνει μια πολύ καλή ευκαιρία συζήτησης και επίσης το ψήφισμα, το εξετάζουμε αυτή τη στιγμή. Τώρα έχετε βεβαίως ανησυχίες για την καθυστέρηση της μεταφοράς του δικαίου. Βεβαίως αυτό είναι θέμα προτεραιότητος και άλλο θέμα που μας απασχολεί είναι η αδυναμία συμμόρφωσης ε, στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ε, η Κομισιόν σε πολλαπλές ε, ανακοινώσεις έχει εξηγήσει πολλές φορές πώς θα πρέπει να εφαρμοστεί το νέο αυτό άρθρο 260 βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας που δημιουργεί καινούρια μέσα. Το έχουμε ήδη εφαρμόσει αυτό, το έχουμε ήδη εξηγήσει στην ανακοίνωσή μας. Έχουμε πολλές περιπτώσεις προσφυγών και πρέπει να δούμε ποιες είναι οι πιο επίγουσες. Γι' αυτό ακριβώς ε, έχουμε ε, καθορίσει μία λίστα προτεραιοτήτων και στην ανακοίνωσή, μου, από το, από το, μας από το 2007 τονίζουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της καθυστερισμένης μεταφοράς του κοινοτικού δικαίου. Ε, και τις συνεπαγόμενες παραβιάσεις. Ιδιαίτερα όταν ένα κράτος μέλος δεν ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τότε θα πρέπει ε, όσον αφορά την εφαρμογή και την μεταφορά του άρθρου 260 της Λισαβόνας. Υπάρχουν, ε, τα ποσοστά που αναφέρεται είναι σωστά. Υπάρχουν όμως και άλλα αριθμητικά στοιχεία τα οποία θα δείχνουν, δείχνουν ότι υπάρχει μείωση των παραβιάσεων και των διαδικασιών προσφυγής λόγω παραβιάσεων σε, από 50% σε 28% περίπου. Ε, οι αριθμοί μπορούν να ερμηνευτούν και διαφορετικά, αλλά βασικά η τάση είναι πτωτική. Όσον αφορά το πρόγραμμα Pilot, το τελευταίο ε, κράτος μέλος που δεν είναι στο pilot είναι το Λουξεμβούργο. Και πιστεύουμε ότι θα καλυφθούν πολύ σύντομα, έτσι ώστε εν τέλει να έχουμε 27 κράτη-μέλη τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα Pilot και καλύπτουν όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα και ελπίζω αυτό να γίνει σύντομα. Όσον αφορά τώρα τα άλλα ε, σημεία που θίξατε, Europe Solve It. Ε, τονίσατε το σημαντικό έργο της Κομισιόν. Το Solve It είναι πραγματικά πολύ επιτυχημένο μέσο. Επιτρέπει την επίλυση κατά 90% των προβλημάτων που θίγουν οι πολίτες μέσα σε ένα διάστημα 10 εβδομάδων, το οποίο είναι ένα πολύ καλό επίτευγμα. Εδώ θα ήθελα να καταλήξω και είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Επειδή προσήλθαν και άλλα μέλη, ρωτώ μήπως έχετε κάτι να προσθέσετε προς το σχόλια. Η κύριε Σιγητά θέλετε να ολοκληρώσετε. Πολύ σύντομα κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που εξέφρασαν την εκτίμησή τους για το σχέδιο γνωμοδότησης. Συμφωνώ με τον κύριο Σβάμπ απόλυτα ότι πρέπει να συνεργαζόμαστε πιο στενά με τα κράτη-μέλη για να τα πείσουμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμόσουν, να μεταφέρουν και να εφαρμόσουν το κοινοτικό δίκαιο. Αυτό το σημαντικό θέμα της συνεργασίας πρέπει να ε, αναπτυχθεί και να ενισχυθεί. Επίσης το Solvit και οι πίνακες συσχετισμών είναι πάρα πολύ σημαντικοί και αναμένω τις τροπολογίες σας για να βελτιώσουμε το κείμενο. Επίσης συμφωνώ με τις δύο συστάσεις της κυρίας Ρούλε και βέβαια χρειάζεται περισσότερη ενημέρωση και βέβαια περισσότερη ε, διαφάνεια αυτό διέπει βεβαίως όλο το κοινοτικό δίκαιο. Ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο της Κομισιόν. It's uh, very good that... Έχω διαπιστώσει όντως ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος και χαίρομαι που η Κομισιόν χρησιμοποιεί ήδη τα μέσα που παρέχει η συνθήκη της Λισαβόνας για να πείσει τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν σωστά την κοινοτική νομοθεσία. Και επίσης είμαι πολύ ικανοποιημένος που το Solvit και το Portal της Europe ε, ε, υποστηρίζεται και ενισχύεται από την Κομισιόν. Αυτή τη στιγμή αναμένω τις τροπολογίες σας και ευχαριστώ όλους τους για τα σχόλιά τους. Η Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Η προθεσμία τροπολογιών είναι 19 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι και θα ψηφίσουμε στο, στην Επιτροπή ΙΜΚΟ 25 Μαΐου. Λοιπόν, ας πάμε στο επόμενο σημείο, καθολικές υπηρεσίες και ο αριθμός ε, εκτάκτου ανάγκης 112. Το σεμινάριο επί του θέματος διεξήχθη πρόσφατα με συνεισφορά εμπειρογνωμόνων διαφόλων φορέων, μη κυβερνητικών οργανώσεων ε, και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον το σεμινάριο και οι περισσότερες παρουσιάσεις έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής μας και να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Σιλβάνα Αράπτη για να μας παρουσιάσει το σχέδιο εκθέσεως. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Το σεμινάριο στο οποίο αναφερθήκατε έγινε χτες το απόγευμα και όντως ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ε, ακούσαμε πάρα πολλές απόψεις και αν μου επιτρέπετε να πω ότι ε, μέσα σε όλη αυτή την κουβέντα που έγινε, ε, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν κοινά σημεία. Και αυτό νομίζω ότι είναι ενθαρρυντικό για την πορεία της υπόθεσης, την πορεία της έκθεσης από εδώ και πέρα και για την πορεία που θα ακολουθήσει ε, μετά την έκθεσή μας και η Κομισιόν. Ε, η έκθεση έχει δύο ε, κομμάτια, αν μπορώ να το πω έτσι. Το ένα αφορά την καθολική υπηρεσία ουσιαστικά και το πλαίσιο των νέων εξελίξεων και το δεύτερο κομμάτι που βεβαίως συνδέεται με κάποιο τρόπο με το, με το πρώτο είναι η υπηρεσία, ο, ο πανευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης 112. Και για αυτό το θέμα έχουμε κάνει μια διεξοδική συζήτηση πριν από ένα-ενάμιση μήνα στην Επιτροπή μας. Τώρα πια ε, έχουμε και ε, το κείμενο στο οποίο κατέληξα ε, λαμβάνοντας υπόψη πρώτον όλη εκείνη τη συζήτηση την πρώτη που είχαμε κάνει στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και βέβαια όπως είπε και ο συνάδελφός μου Μπουσόη στην προηγούμενη έκθεση και όπως ξέρουν όλοι οι συνάδελφοι ε, λαμβάνοντας υπόψη και τον περιορισμό στις λέξεις και την έκταση. Αυτό σημαίνει, και το λέω εκ των προτέρων, ότι με, με πολύ χαρά ε, θα δεχτώ τις απόψεις και τις τροπολογίες των συναδέλφων, όπως επίσης ε, διατυπώνω και τη δική μου πρόθεση να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο το κείμενο ε, σε συνεργασία και με τους ε, σκιώδεις εισηγητές. Δύο κουβέντες, καταρχήν για την καθολική υπηρεσία. Ξέρουμε όλοι ότι από τον καιρό που για πρώτη φορά ορίστηκε η καθολική υπηρεσία, ε, όχι μόνο έχει περάσει πάρα πολύ καιρός, αλλά οι εξελίξεις έχουν τρέξει πάρα πολύ γρήγορα και τρέχουν συνεχώς με αποτέλεσμα να σκεφτόμαστε όλοι πως θα πρέπει να ε, προσεγγίσουμε την καθολική υπηρεσία με έναν άλλο τρόπο. Ε, παράλληλα όμως ξέρουμε όλοι ότι τα ζητήματα αυτά έχουν κόστος έχουμε συνέστηση ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ συγκεκριμένη περίοδο και κοινωνικο-οικονομική πολιτική κατάσταση σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε επίσης στο μυαλό μας ότι το κόστος θέλουμε να επηρεάζει το λιγότερο δυνατό τους Ευρωπαίους πολίτες. Θέλουμε οι Ευρωπαίοι πολίτες δηλαδή να απολαμβάνουν της καθολικής υπηρεσίας σε ποιότητα και ταχύτητα, αλλά να μην επομίζονται δυσβάστακτο κόστος. Αυτά όλα τα λαμβάνουμε υπόψη μας και ξέρουμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε με πολύ προσεκτικά βήματα. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι η καθολική υπηρεσία δεν είναι ούτε δικαίωμα, αλλά ούτε και η βασική όθηση για να πετύχουμε ένα στόχο που λέει ευρυζωνικότητα για όλους. Ο στόχος ευρυζωνικότητα για όλους που αναφέρεται και στο ψηφιακό θυματολόγιο και περιλαμβάνεται στη στρατηγική του 2020, ασφαλώς είναι ένα στόχος τον οποίο υποστηρίζουμε και μάλιστα ένθερμα. Ωστόσο θα πρέπει να τον ζυγίσουμε τον στόχο αυτό, την επιτυχία που θα έχει ο στόχος αυτό σε σχέση με το κόστος. Γι' αυτό και ανέφερα προηγουμένως ότι πρέπει να, να, κάνουμε προσεκτικά ε, βήματα θεωρώ ότι α, η ευρυζωνικότητα για όλους και συνδέω το θέμα αυτό και με το επόμενο κομμάτι της έκθεσης το 112 δεν είναι ο μόνος δρόμος για να βελτιώσουμε ε, την χρησιμότητα, την πρόσβαση και την αποτελεσματικότητα του πανευρωπαϊκού αριθμού κλήσης 112. Υπάρχουν προηγουμένως και άλλα βήματα που θα πρέπει να γίνουν, όπως είναι η συνεργασία των ρυθμιστικών αρχών με τις δημόσιες διοικήσεις, όπως είναι η εφαρμογή τεχνολογιών που ήδη υπάρχουν αλλά δεν χρησιμοποιούνται. Και εδώ πάντα το κόστος είναι, σε σχέση με τους Ευρωπαίους πολίτες, είναι στο μυαλό μας. Κλείνοντας, γιατί δεν θέλω πολύ περισσότερο να ακούσω τους συναδέλφους που ήδη έχουν και το κείμενο και τις πρώτες ε, απόψεις. Ε, θα ήθελα να σας πω ότι και από την χθεσινή ανταλλαγή απόψεων στο σεμινάριο επιβεβαιώθηκε αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, ότι η ευρυζωνικότητα είναι πολύ σημαντικό εργαλείο, αλλά δεν είναι η απόλυτη προτεραιότητα για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Και εδώ έρχομαι και βάζω το θέμα που είναι πάντοτε στο μυαλό μας το θέμα της απόλυτης ε, μέρημνας και φροντίδας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού που οφείλουμε να λαμβάνουμε γι' αυτό μέρημνα και φροντίδα. Ε, από το χτεσινό σεμινάριο πρέπει να πω ότι με ευχαρίστηση είδα πως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβληματίζεται ε, για όλη αυτή την κατάσταση και είναι διατεθειμένη να κάνει ορισμένα βήματα χρήσιμα ε, σε σχέση και με την καθολική υπηρεσία και με τον αριθμό 112 και με την παροχή ευκολιών, διευκολύνσεων στις ευάλωτες ομάδες και ε, στα άτομα με ειδικέ ανάγκες. Εδώ κάπου βάζω εγώ μια τελεία και με πολύ έτσι ανυπομονησία θα έλεγα περιμένω να ακούσω τις απόψεις των συναδέλφων μου. Ευχαριστώ βεβαίως και τους σκιώδεις εισηγητές και τον καλό συνάδελφο κ. Φερνάντες για την εξαιρετική γνωμοδότηση που μας έδωσε πάνω στο θέμα του αριθμού 112 από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Thank you, Madam Σας ευχαριστώ κυρία Ράπτη. Σκιώδης εισηγητής ε, η Ρόζα Γκρίφιν Φόρσταϊν είναι ακόμα καθοδόν για την Επιτροπή. Πάμε στην, επιτροπή, πάμε στην ομάδα Άντε. Λοιπόν, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Αντωνία. Παρα... Κύριε Παρβάνοβα, η συναδελφός μου ζηλεύει γιατί ε, δεν μπορούσε να έρθει εδώ, αλλά ζήτησε να παρουσιάσω την ομιλία της. Θέλω να συγχαρώ εγώ, αλλά και εκ μέρους της κυρίας Παρβάνοβα, την κυρία Ράπτη, για την, ε, το σχέδιο έκθεσης. η προσέγγιση είναι πολύ ισορροπημένη. Δυστυχώς δεν μπορούσα να είμαι παρόν. Στην πολύ καλή, όπως ε, μαθαίνω, στο πολύ καλό σεμινάριο που έγινε χθε το απόγευμα. Αλλά χθε το βράδυ είδα τις παρουσιάσεις, γιατί η γραμματεία του ΙΜΚΟ ε, είχε την καλοσύνη να μας στέλνει τις παρουσιάσεις και ήταν πολύ ενδιαφέρον το σεμινάριο και να συγχαρώ λοιπόν την κυρία Ράπτη για το, το σεμινάριο. Τώρα, α, το σχέδιο έκθεσης, για το σχέδιο έκθεσης ε, έχουμε κάποιες μικρές τροποποιήσεις και προτάσεις. Για την καθολική υπηρεσία είναι, μπορούμε να τονίσουμε ε, δύο έννοιες το θέμα της ε, επικοινωνίας και η ανάγκη της, ε, της ασφάλειας για όλους τους πολίτες. Ε, θα χρειαστεί μια λεπτομερής μελέτη αδικτύπου για το κόστος και την αποτελεσματικότητα για το 112. Χρειάζεται φυσικά η ανάπτυξη τεχνογνωσίας αλλά επίση η αξία και η αποτελεσματικότητα θα πρέπει να αξιολογηθούν από όλου του ενδιαφερόμενου. Μπορεί να λειτουργήσει ο αριθμό, αλλά το θέμα είναι ότι οι υπηρεσίε. Το θέμα είναι τελικά να παρασκευθούν οι υπηρεσίε άμεση ανάγκη το συντομότερο δυνατόν. Ε, θα πρέπει ο χρόνο ε, από την κλήση, από κλήση μέχρι την ε, απάντηση την, ε, να είναι ο συντομότερος δυνατός. Ε, τώρα για το θέμα του αντίστροφου 112 ε, θα μπορέσουν μόνο οι, οι πολίτες που έχουν πρόσβαση στις τηλεπικοινωνίες να έχουν πρόσβαση σε αυτό. Θα, θα πρέπει και αυτό να το αναφέρουμε. Θα χρειαστεί περισσότερο συζήτηση βέβαια, όχι μόνο τις τεχνικές προδιαγραφές και το κόστος, αλλά και για τα, την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Να σας συγχαρώ και πάλι και οι τροπολογίες μας θα έρθουν πολύ σύντομα. Thank you. The next speaker... Επόμενος ομιλητής θα είναι ο Σκιώδης ε, ε, για το, τους πράσινους. Ευχαριστώ λέει η κυρία Ρούλε, και εγώ είχα πάει στην ακρόαση χτες που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Και πολλά ερωτήματα συζητήθηκαν, διευκρινίστηκαν. Βρίσκω την έκθεση αυτή εξαιρετική και αυτά που υπόθηκαν χτες στην ακρόαση αντανακλώνται στην γνωμοδότηση ε, και νομίζω ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε μπορούν να βρουν λύσεις εφικτές. Ε, αυτό που πρέπει να γίνει, κατά τη γνώμη μου, είναι να πιέσουμε την Κομισιόν, να πιέσουμε τη σειρά της η Κομισιόν, τις κρατικές αρχές, να κάνουν πιο ευέλικτες τις, ε, το, κανονιστικό πλαίσιο να το κάνουν πιο ευέλικτο τους κανόνες για τη λειτουργία αυτής της διαδικασίας και να δώσουν τη δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση να δώσει ενισχύσεις να ε, πολλές τοπικές αυτοδιοίκησεις, πολλοί δήμοι φοβούνται να, να, να ξεκινήσουν αυτή τη γραφειοκρατική διαδικασία. Άρα λοιπόν, εφόσον θέλουμε να καλύψουμε και την Ήπεθρο και απομακρυσμένες περιοχές, πρέπει οι κρατικές ενισχύσεις να διέπονται από ένα πλαίσιο αρκετά ευέλικτο, ώστε να μην ε, τρομάζουν τις τοπικές αρχές. Ε, η αναθεώρηση Τις οδηγίες προβλέπει κάτι τέτοιο, αλλά καλό είναι να το τονίσουμε όπου μπορούμε. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. <coughs> Είναι κάποιος από τον που θα ήθελα να σχολιάσει. Και ο εισηγητής ε, από την ομάδα μας ο Σάντορ Αποστέρ δεν είναι εδώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ράπτη και να την ε, συγχαρώ για την εργασία που έχει κάνει. Αντιλαμβάνομαι ότι ο συνάδελφος που παρακολουθεί το θέμα θα υποβάλει τις δικές του εισηγήσει. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα παρακολουθήσουμε το θέμα και θα επανέλθουμε με τον Σάντορ Αποστέρ. Ευχαριστώ πολύ. Διάβασα προσεκτικά τα, τα εγγραφά που ετοίμασε η κυρία Ράπτη και την ευχαριστώ για τη δουλειά της. Ε, συμμετείχαμε και εμείς στην ε, εξαντλητική συζήτηση ε, γιατί θα ήθελα να τονίσω ένα σημείο το οποίο ε, νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε λέτε ότι η καθελική υπηρεσία θα πρέπει να είναι ένα οδηγό ε, για την ευρυζωνικότητα για όλους. Ενώ εγώ πιστεύω ότι καλό θα ήταν να πούμε ότι θα πρέπει να συμπληρώνει όλα τα άλλα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. και τα οποία θα μπορούσαν ε, αυτά να είναι, να είναι οδηγοί. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει μια συμπληρωματικότητα δηλαδή, να έχουμε ευέλικτε λύσει για τα κράτη-μέλη, διότι έχουν διαφορετικέ ε, συνθήκε και θα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι. Ε, και συμφωνώ απόλυτα για το 112 ότι πρέπει να βελτιώσουμε τον το τρόπο εντοπισμού του, του καλούντος και να βελτιώσουμε και την, ε, την ενημέρωση γύρω από αυτό το θέμα. Θα πρέπει οι Ευρωπαίοι πολίτες να γνωρίζουν αυτόν τον αριθμό και να το χρησιμοποιούν και περισσότερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ήρθε ο πρόεδρός μας ο κύριος Χάρμπορ την κατάλληλη στιγμή για να ακούσουμε τα σχόλιά του για το 112. Well, thank you very much, Madam Chairman, and, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, αν έχετε αναρωτηθεί που ήμουν τα τελευταίες 24 ώρες, ήμουνα σε μία αποστολή στο Όσλο, όπου η νοβηγική κυβέρνηση ε, έδειξαν το ενδιαφέρον τους για την εσωτερική αγορά. Για την εσωτερική αγορά. Και απλά αυτό ήθελα να σας ενημερώσω το τι έκανα αλλά παρακολούθησα την ε, έκθεση της κυρία Ζεράπτη, την είχα δει και την προηγούμενη εβδομάδα και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή βάση η έκθεση για την συνεισφορά μας στην ε, διαβούλευση η οποία κάνει αυτή τη στιγμή η Κομισιόν. Νομίζω ότι η κυρία Ράπτη έχει απόλυτο δίκιο στο σχέδιο έκθεσης στο ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτή τη στάση ε, στο να αποφασίσουμε τι θα πρέπει να κάνει το, η Καθολική Υπηρεσία. Νομίζω ότι οι κυβερνήσεις των κρατών έχουν ε, δείξει τη διάθεσή τους να το βάλουν στην μερίσια διάταξη και θέλουν να, να περάσουν σε ένα στάδιο όπου η φρυζενικότητα θα είναι προσβάσιμη σε όλους. Βέβαια η ποιότητα θα ποικίλει ανάλογα με τις περιοχές. Και τώρα το να ε, θέσουμε τεχνολογίες προδιαγραφέ είναι επικίνδυνο. Γιατί η οδηγία για την καθολική υπηρεσία στην οποία ε, ήμουν συγκεκριτή το 2001 και 2002 στη δική μου θητεία στο κοινοβούλιο ε, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι έχουν, οι περιγραφές έχουν κάνει αλματώδη βήματα. Και με βάση την πρώτη δουλειά πλαίσιο ε, έχουν μεταβληθεί πολλά, πολύ τα πράγματα τότε. Η ευρυζωνικότητα έχει αυξηθεί και τώρα έχουμε την ε, επικοινωνία, τη voice communication. Και επίσης έχουν επηρεάσει και το θέμα των κινητών τηλεφώνων έχει επηρεαστεί. Θα ήθελα να προτείνω κάποιες προσθήκες στην έκθεση, ειδικά στο θέμα του, ε, εκεί που τα κράτη-μέλη ε, θέλουν να παρέσχουν ε, ενίσχυση στην ευρυζωνικότητα. Θα πρέπει να δούμε και το θέμα της συμπληρωματικότητας των κινητών και των σταθερών τηλεφώνων. Τώρα για το 1.12. 112. Έχουμε μιλήσει γιατί χαίρομαι που ε, προτείνεται να είναι, γίνει υποχρεωτικά τα e-calls και νομίζω ότι είναι καλή η εποχή για να, ε, να συμμετάσχουμε στη συζήτηση με την Κομισιόν και να μάθουμε το πότε η Κομισιόν θέλει να ολοκληρώσει την ανακεφαλαίωση που κάνουν. Και δεν ξέρω αν αυτό θα συμπεριληφθεί και στην ε, τελική έκθεση της κυρίας Ζεράπτη. Ευχαριστώ. Επόμενη κυρία Περνιού. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστώ την Σιλβάνα Ράπτη για την σύνταξη αυτής της καλής εκθέσεως και για το απόγευμα που διοργάνωσε ε, με όλο το προσωπικό της ΣΥΜΚΟ. Ήταν ένα απόγευμα άκρως ενδιαφέρον για όλους, για όλους τους παρισταμένους και από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και από την πλευρά των διαφόρων μπλεκομένων φορέων όλων όσων ενδιαφέρονται για τις καθολικές υπηρεσίες και για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες. Αυτό που θα ήθελα να πω, έχοντας εργαστεί, έφτασε, ε, έφτασε στην άδεια τώρα που θέλω να μιλήσω, ο Μάλκομ ήρθε τη στιγμή που θα μιλήσω για εκείνον. Ε, συνεργαστήκαμε πολύ, περάσαμε ώρες συζητήσεων επί του πακέτου των τηλεπικοινωνιών και καταφέραμε ε, σε πλήρη αρμονία να εισάγουμε σε αυτό το χαρτοφυλάκιο πολύ σημαντικά στοιχεία για την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών κυρίως ε, τα, τα, για τα ευάλωτα άτομα και τα άτομα με αναπηρία. Ε, είναι καλό που βρίσκουμε αυτά τα στοιχεία εδώ. Μπορούμε να συζητήσουμε εκτενώς κατά πόσο οι καθολικές υπηρεσίες είναι δικαίωμα ή όχι. Είναι στον αριθμό 6 της εκθέσεως της ε, Σιλβάνας. Εν πάση περιπτώσει η πρόσβαση σε μια καθολική υπηρεσία, σε ποιοτικές καθολικές υπηρεσίες σε ανεκτή τιμή θα πρέπει να είναι για μας ένας στόχος προς επίτευξη. Έχουμε μέσα στα πλαίσια της συνθήκης της Αβώνας έχουμε όραμα και στόχο την κοινωνική συνοχή και την εδαφική συνοχή. Αυτό είναι σημαντικό. Ε, έχουμε επίσης και τη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων για τους πολίτες. Νομίζω ότι με αυτά τα δύο μέσα, τα εργαλεία αυτά, μπορούμε να κερδίσουμε την πορεία μας, που είναι σημαντικό αυτό αν θέλουμε να ε, σταματήσουμε τον κατακαιρματισμό που υπάρχει. Κυρίως και τη διαφορά, το ψηφιακό χάσμα. Ε, ευρυζωνική είναι δυνατή για όλους. Όχι, αμέσως χρειάζονται πολλές επενδύσεις, μεγάλες επενδύσεις, πρέπει να γίνουν σοβαρές αξιολογήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφωνώ με την κυρία Ρούλε, θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τις τρευλώσει του ανταγωνισμού, αλλά όσον αφορά το 112, είναι για κατεπίγουσες κλήσεις αυτός ο αριθμός. Ταυτόχρονα Όμω είναι περισσότερο μια υποχρέωση που έχει η Ευρώπη έναντι των πολιτών, διότι αφορά την υγεία του, αφορά την ασφάλεια τη ζωή του, είναι κάτι πολύ θεμελιώδε και θα πρέπει πραγματικά να επιταχύνουμε τη διαδικασία και εδώ θα πρέπει ο καθένα να υπομειστεί τι ευθύνε του. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ του και οι διάφορε εταιρείε Όταν μιλάμε για επενδύσει, να μην λησμονούμε ότι υπάρχει πάροχοι ε, εμπλέκονται και σε περίοδο οικονομικής κρίσης ε, θα πρέπει ε, κάνουν κέρδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βγάζουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Θα πρέπει εν μέρη τα κέρδη να επενδυθούν σε υπηρεσίες προς πολίτες όπως το 112. Και για το 112 το συζητήσαμε εκτενώς. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ζήτησα χτες από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δράσει λέγω Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ίδια συναρτήσει των δυνατήτων που τις παρέχουν οι αρμοδιότητές της για να πιέσει τα κράτη-μέλη να ευαισθητοποιήσουν καλύτερα τον κόσμο για το 112. Είναι σημαντικό. Στη χώρα μου το 112 είναι σχεδόν άγνωστο. Ε, χτες μιλήσαμε 26% και εξεπλάγει χτες τα άκουσα. Ε, και ο γεωλογικός εντοπισμός είναι, ε, ο γεωγραφικός εντοπισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Πρέπει να υπάρχει ε, η πολιτική βούληση, το μπαλάκι είναι στο γήπεδο του Κοινοβουλίου, είναι πιο προχωρημένο στις συζητήσεις και στον προβληματισμό το Κοινοβούλιο και τα Κοινοβούλια ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν πιέσουν τα κάτι μελη μπορούμε να προχωρήσουμε σχετικά ε, γρήγορα και να κάνουμε κάτι στους πολίτες. Σας ευχαριστώ, Σιλβάνα. Ευχαριστώ. Άλλος, ο οποίος θέλει να σχολιάσει, αν δεν υπάρχει άλλος, θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Ράπτη. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Παρακολουθώντας την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έγινε τα προηγούμενα λεπτά, ε, έχω να σημειώσω τα εξής. Πρώτον, ε, ήξερα, αλλά βλέπω και ακούω με πάρα πολύ χαρά αυτή την εξαιρετική συνεργασία που υπήρχε μεταξύ του συναδέλφου κυρίου Χάρμπορ και της συναδέλφου της κυρίας Μπερναντέτ Βερνιό και είναι κατά κάποιο τρόπο τους νιώθω σαν τον πατέρα και τη μητέρα αυτού του δεκάχρονου παιδιού που παραλαμβάνω εγώ σήμερα. Ε, οι παρατηρήσεις τους ε, είναι πάρα πολύ εύστοχες και με βάζουν σε έναν πολύ θετικό προβληματισμό. Ε, συμφωνώ συμφωνώ και με τις παρατηρήσεις που έκανε ο κύριος Χάρμπορ και με τις επισημάνσεις της Περναντέτ και τους ευχαριστώ. Ο συνάδελφος κύριος Μπουσόη ε, ανέφερε τρία ζητήματα τα οποία με απασχολούν και ευχαριστώ που βλέπω να έχουμε συμφωνία μιλάω για το χρόνο ανταπόκρισης, μιλάω για τον εντοπισμό του καλούντος και μιλάω και για το αντίστροφο 112. Ε, σημειώνω εδώ ότι η κυρία Παρβάνοβα πέρασε εκτές ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από την ακρόαση που είχαμε από το σεμινάριο και την ευχαριστώ γι' αυτό, όπως ευχαριστώ και τον κύριο Μπουσό για τις ε, ε, επισημάνσεις του. Και σε σχέση με τον εντοπισμό ε, πάω αμέσως και θα καταλάβετε γιατί, στις παρατηρήσεις της Ρόζας που α, ήταν χτες όλο το σεμινάριο και επίσης την ευχαριστώ που όλο του το απόγευμα ήταν εδώ. Ε, μας είπε ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα χτες το βράδυ που αξίζει να το επαναλάβω νομίζω όταν οδηγούσε κάπου στην Γερμανία και μέσα στη νύχτα α, βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν αγριόχειρο Έκανε λοιπόν τηλεφώνημα στο 112, όπου όμως υπήρχε δυσκολία να την εντοπίσουν. Ο λόγος ήταν ότι ήθελε να προειδοποιήσει και τους άλλους οδηγούς που ήταν στον αυτοκινητόδρομο ότι υπάρχει αυτό το γεγονός εκεί. Είναι ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα που μας κάνει ε, ακόμη περισσότερο να συνειδητοποιούμε πόση ανάγκη υπάρχει για να μπορεί να γίνεται ο εντοπισμός του καλούντος. Ε, τώρα, η Ρόζα έθεσε και ένα άλλο σημείο σε σχέση με την ευρυζωνικότητα. Ε, το έψαχνα εδώ τα χαρτιά μου και είναι ακριβώς στο σημείο 6 που στην ελληνική μετάφραση που έχω μπροστά μου είναι ότι η καθολική υπηρεσία, ότι η ευρυζωνικότητα για όλους δεν είναι, πώς να το πω, αυτοσκοπός, δεν είναι ε, ε, ε, ένα θέμα από μόνο του. Είναι ασφαλώς να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τα υπόλοιπα, όπως το είπε η Ρόζα. Ε, απλώς ανέφερα στην εισήγησή μου και χτες και την προηγούμενη κουβέντα που είχαμε κάνει ότι η ευρυζωνικότητα ως στόχος έτσι όπως περιγράφεται στην στρατηγική της Ευρώπης 2020 στην ψηφιακή ατζέντα πάντα υπάρχει στο μυαλό μας. Αλλά ασφαλώς η συμπληρωματικότητα ε, είναι στην, ε, στη ζωή μας. Ευχαριστώ τον Κυριάκο Τριανταφυλλίδη που εξέφρασε τη διάθεση και τη δική του εκπροσωπώντας και τον σκιώδη συγητή της ομάδας του. Ε, ξεχνάω κάτι, αν ξεχνάω να με βοηθήσετε κυρία Πρόεδρε. Ε, και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που είναι εδώ, που άκουσαν και που με πολύ χαρά θα δεχτώ τις τροπολογίες τους, τις υποδείξεις τους, τις παρατηρήσεις τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Φαντάζομαι δεν ξεχάσατε τίποτα. Πρώτον, αυτό είναι καλό. Σημαίνει ότι λειτουργεί καλά εδώ το μυαλό. Ε, ξέχασα όμως, τώρα θυμήθηκα τι ξέχασα να πω, ε, μου δημιούργησε μία ε, αισιοδοξία η τοποθέτηση και η στάση την οποία κράτησε χτες στο σεμινάριο ο εκπρόσωπος της ε, Κομισιόν, ο κύριος Λάιχαν, αν σωστά το προφέρω, αυτό το όνομα το στραμπούληξα λιγάκι, ε, ο οποίος πραγματικά μας άφησε να ένα περιθώριο να ελπίζουμε ότι ε, και η Κομισιόν έχει αντιληφθεί πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Και αυτό θεωρώ ότι είναι θετικό για τους Ευρωπαίους πολίτες. Excellent. Um, Έξοχα. Να σας θυμίσω την προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. 18 Απριλίου στις 6 το απόγευμα. Καλώς. Πάμε στο σημείο 7, κύριε Πρόεδρε. Κανείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι. Κύριε Χάρμπορ, θέλετε να συνεχίσετε. Θα συνεχίσω λοιπόν εγώ, όσο παίζει το ρόλο του σκιώδου συζητητού, το σημείο 7, πιο αποδοτική, πιο αποτελεσματική και δίκαια αγορά λιανικής. Η κυρία Άννα Μαρία Κοράτσα, α, δεν είναι εδώ, είναι καθοδόν. Θέλετε να μας πείτε για την επίσκεψή σας στο Όσλο. Αν συμφωνούν οι συνάδελφοι, ώσπου να έρθει η κυρία Κοράτσο Μπίλτ, η κυρία Ράπτη τα ολοκλήρωσε πάρα πολύ ωραία. Θα μπορούσα να μιλήσω. Καλό θα ήταν να είχαμε ακούσει για την έρευνα που έχει γίνει μέχρι τώρα, διότι όπως ξέρετε έγινε μια διαδικασία διαβούλευσης και η Κομισιόν τώρα εξετάζει τα συμπεράσματα αυτής της διαδικασίας και πριν κάνει μια, πριν κάνει μια επίσημη πρόταση το φθινόπωρο για την επίσκεψή μου στην Ορβηγία. Ο λόγος για τον οποίο πήγα στην Ορβηγία είναι επειδή η Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ε, είχε οργανώσει μία συνάντηση ταυτόχρονα και μπόρεσα έτσι να εκμεταλλευθώ την διοργάνωση αυτή. Η κυρία Στέλλερ με συνόδευσε σε όλες μου τις συναντήσεις και αυτό ήταν πάρα πολύ χρήσιμο, η παρουσία της δηλαδή, και ε, η ΙΜΚΟ ε, εκπροσωπήθηκε και ο κύριος Τσαρκόφσκι ο οποίος όπως ξέρετε κάνει μια έκθεση πρωτοβουλίας για την εσωτερική αγορά και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, τον ΕΟΧ. Αυτή η έκθεση ε, σε, ακόμα εκτιμάται ιδιαίτερα, ε, είναι επίκαιρη και ε, στη συνάντηση αυτή τονίστηκαν τα σημαντικά οικονομικά θέματα της Ένωσης και του ΕΟΧ από τους εταίρους. Εχθές το πρωί είχα μια συνάντηση προγεύματος με τον Νορβηγικό Σύνδεσμο Βιομηχανιών και εν συνεχεία συνάντηση με τον Υπουργό Βιομηχανίας. Εν συνεχεία συνάντησα δύο υπουργού υπεύθυνου για τις δημόσιες προμήθειες και την προστασία των καταναλωτών. Και Τέλος, ε, μας ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Είχαμε ένα briefing. Ε, πολύ, λοιπόν, ε, δραστήρια μέρα. Τώρα, για την εσωτερική αγορά μπορώ να σας πω ότι οι Νορβηγοί υποστηρίζουν έντονα τη συμμετοχή τους στην εσωτερική αγορά. Αν δείτε το βαθμολόγιο της εσωτερικής αγοράς, θέμα της κυρίας Τούν, θα δείτε ότι το έλλειμμα μεταφοράς δικαίου είναι το μικρότερο στην Νορβηγία. Δηλαδή έχουν την καλύτερη βεσμολογία στο θέμα της μεταφοράς δικαίου, κανονισμών κλπ. από όλες τις άλλες χώρες. Την καλύτερη βασμολογία για την εφαρμογή της νομοθεσίας. Ιδιαίτερα στις δημόσιες προμήθειες, η Νορβηγική Υπηρεσία Δημοσίων Προμηθειών, που συνδέεται με την Επιτροπή Ανταγωνισμού παρακολουθεί πολύ προσεκτικά τις όλες ε, τις διαδικασίες δημοσίων μειοδοτικών διαγωνισμών έτσι ώστε να είναι συμβατές με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αλλά ταυτόχρονα επιδιώκει καινοτομικές ε, λύσεις και διαδικασίες. Αυτή η δημόσια υπηρεσία προμηθειών είναι πάρα πολύ χρήσιμη και επικοδομητική και καλό θα ήταν να την καλέσουμε σε μία μελλοντική ακρόαση. Θα ήταν πραγματικά πολύτιμη η συμβολή των Νορβηγών εμπειρογνωμόνων. Έχουμε πάρα πολλά να μάθουμε από αυτούς. Όταν συναντήθηκα με τον Υπουργό Προστασίας Καταναλωτών, με την Υπουργό και κοινωνικής ενσωμάτωσης ε, ασχολείται ιδιαίτερα με την παρακολούθηση της πράσινης πτυχής στις δημόσιες ε, προμήθειες και στα θέματα προστασίας των καταναλωτών. Δηλαδή θέματα που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Στα θέματα των καταναλωτών ε, ακούσαμε ορισμένες επιφυλάξεις των Ορβηγών όσον αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών, ε, ορισμένες επιφυλάξεις ε, στις τρέχουσες προτάσεις που προέρχονται από μας. Ιδιαίτερα για την οδηγία του Συμβουλίου, η οποία ενθαρρύνει το ελάχιστο επίπεδο προστασίας καταναλωτών. Ε, όμως τόνισαν ιδιαίτερα τα συστήματα ADR, δηλαδή συστήματα απάλληψης διακρίσεων ανάλογα με το γένος και έχουν μία εξαιρετικά δραστήρια Επιτροπή Ισότητος και Προστασίας Καταναλωτών. Μπορούμε λοιπόν να εξετάσουμε τις δικές τους διαδικασίες σε βάθος όταν θα έχουμε στα χέρια μας την επόμενη έκθεση της Κομισιόν για αυτά τα θέματα. Ο Υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας επίσης εξέφρασε την ε, θερμή του υποστήριξη για την εργασία που κάνουμε στα θέματα της εσωτερικής αγοράς και μου ε, τόνισε ε, την υποστήριξη της κυβέρνησης σε όλα τα θέματα της εσωτερικής αγοράς. Οπότε με την ευκαιρία αυτή τον κάλεσα να έρθει σε μας και να μιλήσει την Επιτροπή μας. Πιστεύω ότι και εσείς θα θέλατε να το γνωρίσετε και να ακούσετε τι έχει να μας πει ο Υπουργό ε, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Θα το κανονίσω λοιπόν τις επόμενες έξι μήνες. Τι έχει να μας πει για την κοινή αγορά. Και τέλος, ε, αυτή τη στιγμή εκπονούν, εκπονείται μία μελέτη ε, από πλευράς Νορβηγίας, την οποία έχουν αναθέσει σε ένα σώμα ακαδημαϊκών εμπειρογνωμόνων για το μέλλον των συμφωνιών ε, μεταξύ Νορβηγίας και των άλλων ε, χωρών του ΕΟΧ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, είναι μία μελέτη η οποία θα εξετάσει το ακίκο το κοινοτικό και εκτιμένο, το παλαιότερο, το οποίο βασιζόταν κυρίως στους πυλώνες και τις νέες εξελίξεις ε, με τη νέα συνθήκη στα θέματα της ε, κοινή ε, και εσωτερικής αγοράς. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι Στη Νορβηγία συζητώνται έντονα τα, οι εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή την εξουσία την έχει το Εργατικό Κόμμα και η διάσκεψη, το συνέδριο του Εργατικού Κόμματος πρότεινε να συνυπογράψει η Νορβηγία την τρίτη οδηγία, ε, ταχυδρομική οδηγία. Την τρίτη οδηγία για τα ταχυδρομεία. Ε, και αυτή τη στιγμή διενεργεί μια εκστρατεία για να πείσει τους, ευρω... τους νορβηγούς ψηφοφόρους ε, για τα ωφέλη τα οποία θα προκύψουν από αυτήν την ε, συμμετοχή. Ήμουν πολύ ευτυχής που είχα την κυρία Στάιλερ μαζί μου να με συνοδεύει, εκπροσωπήσαμε την ΙΜΚΟ και παρουσιάσαμε τις θέσεις μας και πιστεύω να συμφωνείτε ότι είναι σωστή η πολιτική αυτή της Επιτροπής μας να συζητούμε με την νορβηγική κυβέρνηση, με τους νορβηγούς συναδέλφους, διότι η συμμετοχή και η υποστήριξή τους στην εσωτερική αγορά είναι έντονη, πολύ σημαντική. Μπορούμε να επανέλθουμε τώρα στην έκθεση για πιο αποτελεσματικό και δίκαιο λιονεμπόριο. Να δώσω το λόγο στη συγκεντρία Κορατσαμπίλτ. Χαίρομαι πολύ ε, που φτάσαμε στη σημερινή μέρα. Ε, είναι πολύ σημαντική για μένα. Ε, ασχολούμαι με πολλές... Είναι η πρώτη δική μου έκθεση ως εισηγήτρια. Έχω εδώ μία μάδα φοιτητών από τη Σουηδία που μας επισκέπτονται και θα ήθελα να τους καλωσορίσουμε. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι αυτή η έκθεση ξεκινά να συζητείται ε, αμέσως μετά το ψήφισμα ε, του νόμου για την εσωτερική αγορά. Ε, έχουμε ανάγκη από μια πιο λειτουργική εσωτερική αγορά και γι' αυτό νομίζω ότι δεν επαναλαμβανόμαστε γιατί το, το λιανική αγορά είναι πυλώνας της εταιρική αγοράς. Εδώ πέρα πρέπει να αναφέρουμε όλους τους ενδιαφερόμενους και την αλυσίδα εφοδιασμού και τους λιανεμπόρους. Δεν μπορούμε βέβαια στις λίγες σελίδε να τους αναφέρουμε παντού, αλλά πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η διάσταση Σούμαν. Είναι η ανθρώπινη διάσταση λοιπόν. Γι' αυτό και μιλάω και για ευέλικτες δουλειές. Flexible jobs. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ καιρό αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας και έχουν την ευκαιρία να επανέλθουν. Ανθρώπους που έχουν λιγότερους ευκαιρίες για σπουδές, αλλά και ε, ανθρώπους που δουλεύουν στην υψηλή τεχνολογία. Οπότε ε, μιλάμε για πολλές, ε, πολλά επίπεδα. Μιλάμε για ανθρώπους από άλλες χώρες, για τις γυναίκες και δίνεται η δυνατότητα να εργαστούμε ανάλογα με τις απαιτήσεις σύγχρονης ζωής. Ένα άλλο ζήτημα, η ποικιλία στην προσφορά των καταναλωτικών αγωθών. Ο καταλύτης θέλει αυτή ποικιλία. Για μένα λοιπόν η λέξη ευελιξία είναι η πιο θετική που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω για να περιγράψω τον τρόπο που η λιανική αγορά δίνει ευκαιρίες. Μαζί με την ε, σκιώδη μου εισηγήτρια, ε, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω και να ξαναδουλέψω μαζί του. Είμαστε υποχρεωμένοι να επικεντρωθούμε και να βάλουμε προτεραιότητες σε αυτή την έκθεση. Ε, δεν είναι μία έκθεση που αφορά συγκεκριμένα την εργασία ή κάτι άλλο, αλλά έχουμε επικεντρωθεί στο θέματα καθαρά εσωτερικής αγοράς. Έχουμε εντοπίσει τέσσερι ε, τομείς όπου χρειάστηκε να δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα. Και προσπαθήσα, προσπαθήσαμε να, να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Δεν, ε, η προσέγγιση μου δεν ήταν ιδεολογική, αλλά πραγματιστική ε, εταιρείες όπως η Coca-Cola έχουν ε, χαλάσει τη σχέση τους. Η Coca-Cola πλέον δεν πουλάει π.χ. για το, τη συσκευασία ενός λίτρου στο ΙΚΑ. Και αυτό μπορεί να μας δείξει το πώς μπορεί να οι πολίτες να ασκήσουν την ελευθερία επιλογής στο κατανάλωση και να επηρεάσουν ε, την κατάσταση. Ένα άλλο θέμα, ελευθερία κινήσεως. η ελευθερία ε, κινήσεως των αγαθών. Παντού έχουμε πάλι μια συγκεκριμένη α, προσέγγιση και χρειαζόμαστε συγκεκριμένες λύσεις. Για μένα ε, είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε περιοριστικά ε, εθνικ, περιοριστικούς εθνικούς κανόνες όπως ε, ε, κανόνες πιστοποίησης και το θέμα είναι να εφαρμόζεται σωστά η νομοθεσία για την εσωτερική αγορά. Έχουμε τα εξαιρετικά μέσα όπως το Solvit και το IMI και το σύστημα πληρωμών ε, είναι προβληματικό για την ελεύθερη διακίνηση των αγαθών και θα ζητήσω με την Κομισιόν να, να, ε, να θεωρήσει το σύστημα ΣΕΠΑ ε, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληρωμών και να καταργήσει έτσι ε, τα επιπλέον ε, τέλη τα οποία υποχρεώνεται να πληρώσει κανείς. Ένα άλλο θέμα. Έχουμε ανθρώπους που ζουν στην Ήπεθρο, στην πόλη. Όλοι έχουν το δικαίωμα ίσες πρόσβαση στην αγορά. Όπως και οι επιχειρήσεις θα είχαν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση ε, σε ολόκληρη την αγορά. Στην, στον, ο νόμος για την ενιαία αγορά, για την κοινή αγορά θα πρέπει να ε, ε επιβληθεί. Το e-commerce τώρα, το ηλεκτρονικό εμπόριο, είναι πολύ σημαντικό για μας και ζητάμε να χτίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών προς, αυτό, το ηλεκτρονικό εμπόριο δηλαδή. Το θέμα το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν είναι ανταγωνιστικό προς το κανονικό εμπόριο, απλά είναι συμπληρωματικό. Το πιο... το πιο δύσκολο σημείο είναι το... οι σημαντικές σχέσεις. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ε, ή ότι η σύγκρουση που υπάρχει αυτή τη στιγμή ότι είναι επικοδομητική. Υπάρχουν εμένα προβλήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ε, όμως σε ένα πιο σωστό κλίμα. Να χτίσουμε τις σχέσεις εμπιστοσύνης, να περάσουμε από μια σχέση σύγκρουσης σε μια ε, σχέση επικοδηματικού διαλόγου και άμεσου διαλόγου. Δεν νομίζω ότι μικροδιαχείριση θα βοηθούσε. Το καλύτερο που μπορεί να κάνει το κοινοβούλιο είναι να διευκολύνει τη διαδικασία μεταξύ των ενδιαφερομένων α, να λύσουν μεταξύ τους τα προβλήματα. Με την ε, ε, βοήθεια φυσικά της Κομισιόν, σαν ανεξάρτητο ε, σώμα, το οποίο θα μπορούσε να, η οποία Κομισιόν θα μπορούσε να βοηθήσει. Να περάσει το, να περάσουμε από μια κατάσταση σύγκρουσης προς μια πιο επικοδοματική σχέση. Γι' αυτό θα θέλαμε να μας βοηθήσει η Κομισιό να, να εντοπίσουμε ποιες εμπορικές πρακτικές είναι άδικες, για παράδειγμα. Ποιες είναι μη ανταγωνιστικές πρακτικές ή και παράνομες πρακτικές στο εμπόριο. Ε, βέβαια πρέπει να υπάρξει με καλύτερη εφαρμογή του δικαίου της ανταγωνιστικότητας και σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Να εξεταστούν οι βέλτιστες πρακτικές. Πώς εφαρμόζεται το δικαίωμα ανταγωνισμού και να δώσουμε μια προθεσμία μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς για να έχουμε μια πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα της κατάστασης για να δούμε πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε αφήνω ανοιχτά κάποια θέματα κυρία Πρόεδρε, διότι στο θέμα των συμβατικών σχέσεων στο φόρουμ υψηλού επίπεδου, είναι σε έξι μήνες και πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία σε αυτές τις πλατφόρμες να εκδηλώσουν κάποιες τάσεις πριν να τις προκαταλάβουμε εμείς. Προτείνω τρεις επιλογές που βέβαια μπορεί να προτείνουν και να να προτεθούν και άλλες επιλογές. Να ενδυναμώσουμε την ε, συζήτηση στην υπάρχουσα πλατφόρμα ε, ή να ακολουθήσουμε την πρωτοβολία που ο επιχειρηματικό κόσμος έχει ήδη ξεκινήσει. Θα ήθελα οι συνάδελφοι να ακούσουν ότι ο επιχειρηματικός κλάδος, οι λιανέμποροι λαμβάνουν ήδη βήματα τα οποία εγώ τα θεωρώ σημαντικά, δείχνουν μια προθυμία να μιλήσουν και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Ε, περάσαμε από το στάδιο της άρνησης ότι υπάρχουν προβλήματα και πλέον έχουμε περάσει σε ένα στάδιο ο, του να μπούμε σε φόρα όπως το Eurocommerce και άλλα όπου εκεί υπάρχει η διάθεση να κάτσουμε στο τραπέζι με την Κομισιόν. Δεν έχουμε δει ακόμα τεράστια αποτελέσματα, αλλά η διαδικασία έχει ξεκινήσει και εμείς θα πρέπει να την ενισχύσουμε. Η τρίτη επιλογή είναι ε, το να, η δημιουργία ενός νέου φόρουμ με λιγότερη, μεγαλύτερη εστίαση στο, στα κλάδα των τροφίμων αλλά να έχει ένα πιο ευρύ πεδίο εφαρμογή. Και κάθε τέτοια πρωτοβουλία, κατά τη γνώμη μου, αν είναι, κινείται προ τη κατεύθυνση, θα πρέπει να την ενισχύσουμε. Βέβαια, υπάρχουν και άλλε επιλογέ που θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη μα. Και θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε αυτές. Προτείνω μια, ετήσια, ένα, μια στρογγυλή τράπεζα για το λιανεμπόριο, όπου θα μπορούμε να δούμε τι έχει ήδη επιτευχθεί και άλλες προτάσεις. Ας μην κλείσουμε την πόρτα, ας δώσουμε ευκαιρία στο διάλογο να δώσει τα δικούς του καρπούς. Άλλο σημαντικό σημείο είναι η βιώσιμη κατανάλωση. Οι καταναλωτικές οργανώσεις πραγματικά μας έχουν ζητήσει να το δούμε αυτό. Και το λιανεμπόριο έχει τεράστια ευθύνη όσον αφορά την οργάνωση, τις μεταφορές με πιο βιώσιμο τρόπο, τη διαχείριση των αποβλήτων και θα πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία να μας δείξουν ε, τα, το τι έχουν κάνει τι έχουν ε, επιτύχει, που οι πολίτε μπορεί να μην το γνωρίζουν. Τέλο, κοινωνικό διάλογο. Ο κοινωνικό διάλογο μπορεί να μην λειτουργεί σωστά στο κλάδο του εμπορίου. Εγώ τουλάχιστον έτσι νομίζω. Είναι ένα παράδειγμα όπου. Α, όχι, ε, ε, έχει λειτουργήσει μάλλον σε αυτό το κλάδο. Και το Eurocorments και το Uni Europa έχουν, ε, έχουν κάνει πολύ καλές πρωτοβουλίες και θέλω και να τους συγχαρούμε γιατί μπόρεσαν να χτίσουν το, τη συνένεση. Οπότε εδώ δεν ότι δεν χρειάζεται να επέμβουμε. Ας τους υποστηρίξουμε ε, στη μάχη τους για μείωση ε, της ε, της εργασίας στον τρόπο που ενισχύουν την εταιρική ευθύνη και άλλα μέτρα που προτείνουν σαν φορείς. Επειδή το κλάδος του λιανεμπορίου είναι τόσο σημαντικός και επειδή υπάρχουν τόσες πολλές προκλήσεις, νομίζω ότι χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση. Να ζητήσουμε και από την Κομισιόν να πάρει μια τέτοια ολιστική προσέγγιση και να ζητήσουμε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράση για το λιανικό εμπόριο. Αυτό θα μπορούσε να ε, ενισχύσει τις προσπάθειές μας μακροπρόθεσμα Έχουμε ήδη ψηφίσει ε, μια τέτοια πρόταση, ένα τέτοιο μέτρο στον ε, νομοθεσία για την ενιαία κοινή αγορά και θα ήθελα να ακούσω και τις δικές σας ερωτήσεις και τις δικές σας ε, συνεισφορές. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Κόρατσα Μπίλτ. Λοιπόν, θα ήθελα να καλωσορίσω φοιτητές από τη Σουηδία που είναι εδώ και να σας πω ότι μπορείτε να είστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για όλους τους Σουηδούς βουλευτές που είναι παρόντες εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά λοιπόν και θα πάμε στον επόμενο μιλητή, σκιώδης εισηγητής από τη σοσιαλιστική ομάδα, η κυρία Παντζέρη. Ο κύριος Παντζέρη, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια καταρχάς για την συνεργασία μας αυτούς τους μήνες και στις συναντήσεις που κάναμε εδώ στις Βρυξέλλες και σε αυτές που έλαβαν χώρα στο Στρασβούργο. Είναι πολλά τα σημεία επί των ομοίων ε, συζητήσαμε και υπογραμμίσαμε τα σημεία, δεν μπορώ να τα παριθμίσω όλα, αλλά θα τονίσω την, την ανάγκη να αρθούν τα εμπόδια που εμποδίζουν σε αυτό το τομέα την επίτευξη του πλήρους δυναμικού του και σε αυτό το πλαίσιο χρειάζεται να εφαρμοστεί επαρκώς η ισχύουσα νομοθεσία. Ε, πιστεύω μετά ότι χρειάζεται να υποστηρίξουμε τις συμφωνίες με το, το, το, των κοινωνικών και τον κοινωνικό διάλογο. Χρειάζεται ευρωπαϊκό σχέδιο ω σφαιρικό για το λιανεμπόριο για να αντιμετωπίσουν τα ανεπίλητα ζητήματα και να μπορούν να δοθούν ίσως και συστάσεις συγκεκριμένες για κάθε τομέα. Η συγγήτρια νομίζω σωστά αναφέρθηκε στην ανάγκη μιας ολιστικής προσέγγισης που θα ενισχύσει το συντονισμό των διαφόρων πολιτικών. Πρόκειται περιουσιαστική σημαντικής πτυχής. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο πιστεύω ότι τα πολλά θέματα που ήδη εφήχθησαν στην έκθεση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και τις πτυχές από οποίων χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή, κυρίως για να δοθεί συνοχή και συστηματική προσέγγιση στην ε, έκθεση συμπερίληψη που θα εμπλουτίσουν τη σημαντική εργασία που ετεύχθη και πάνω σε αυτό θα αναφέρω τέσσερα σημεία. Ε, το πρώτο σημείο. Πρέπει να εστιαστούμε περισσότερο επί των καταναλωτών και της εφαρμογής των προδιαγραφών για τα κοινωνικά δικαιώματα και για την εργασία. Πικίλη νομοθεσία από χώρα σε χώρα όσον αφορά αυτά τα θέματα. Δεύτερο σημείο, αφορά την ανάγκη να υπογραμμίσουμε ότι η βελτίωση των συνθήκων εργασίας, η καταπολέμηση της μαύρης οικονομίας και η διατήρηση του πεπέδου απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας μέσω καλύτερης ανταπόκρισης της ανάγκης των εμπόρων και των εργαζομένων είναι οι βασικές προκλήσεις σε αυτό το πεδίο. Αυτές είναι ενδείξεις που ήδη παρουσιάζονται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα πρέπει να ενισχύσει και η αρμοδιότητα της Επιτροπής μας. Θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην έκθεσή μας ε, για να κινηθούμε με ολιστικό πνεύμα όπως αναφέρθηκε όσον αφορά την προβλημάτων. Το τρίτο που θα ήθελα να θίξω, θα πρέπει να αναφέρουμε και μια ευρύτερη έννοια της ευθύνη των επιχειρήσεων. Δηλαδή, κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη που συμπεριλαμβάνονται για την επιχείρηση, ευθύνη επιχείρηση. Και τέταρτον, θα πρέπει να ίσω να υπογραμμίσουμε το ρόλο των συνεταιρισμών στο σύστημα τη διανομή των εμπορευμάτων στη Λιανική, διότι αποτελούν ένα εναλλακτικό εμπορικό σύστημα που συμβάλλει στον οικονομικό πλουραλισμό, που δίνει πρόσβαση, ε, καλές τιμέ, ποιότητα και υποστηρίζει και την τοπική παραγωγή Αυτέ είναι κάποιε προτάσει, κάποιε συστάσει, κάποιε ενδείξει που πιστεύω ότι ήταν χρήσιμε να ενταχθούν για να εμπλουτίσουν μια έκθεση που, όπω είπα, είναι πολύ σημαντική. Και ευχαριστώ εκ νέου για αυτό την εισηγήτρια, για την προσπάθεια που έκανε. Και είναι σημεία που, πώ να το πω, θα βρουν πλήρη αναφορά, πλήρη εξήγηση σε τροπολογίε. Και εύχομαι μετά να υποστηριχθούν οι τροπολογίε μου και από την εισηγήτρια και από όλη την Επιτροπή. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την άποψή μου σχετικά με αυτή την ε, έκθεση. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Ρε Πρόεδρος. Σκιώδης της Άλντε θα αντικατασταθεί από τον κύριο Κρόιτσμαν. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ο κύριο Λέντεργκάρ θα ήθελα ευχαριστήσει την εισηγήτρια για μια ανοιχτή διαδικασία με μεγάλη συνεργασία και μια πάρα πολύ καλή έκθεση. Και οι παραγωγοί και οι λιανοπολιτέ φοβούνται ότι θα ήταν μη ισορροπημένη και μεροληπτική έκθεση. Ο κ. Γέρεγκαρτ πιστεύει ότι η ισορροπία του κειμένου έχει επιτευχθεί λίγο πολύ. Ήταν ζωτικό για τον κ. Λίδεγκαρτ να τονιστεί η ανάγκη για σωστή εφαρμογή και επιβολή της σα νομοθεσία για την εσωτερική αγορά. Αυτό είναι κάτι που συμπεριλαμβάνεται. Επίση, ήταν ζωτικό για τον κύριο Λίντεγκαρτ να μην καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίζει νομοθεσία για άδει, εμπορικέ πολιτικέ, αλλά να κληθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει αξιολόγηση συνεπειών πριν προχωρήσουμε περαιτέρω. Ο κ. Ζέντεγκαρντ θα υποβάλει κάποιε τροπολογίε για το κείμενο, αλλά όχι κάτι, δεν θα προτείνει κάτι που θα αλλάξει εξ ολοκλήρου την ισορροπία. Αυτά και ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Η ε, κυρία Ρούλε. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαιρετική συνεργασία. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές μαζί και γενικά νομίζω ότι η έκθεσή σας ε, συμπεριλαμβάνει, καλύπτει τα βασικά προβλήματα. Αλλά βεβαίως η αηφόρος κατανάλωση πιστεύω δεν καλύπτεται επαρκώς. Πρέπει να προσέξουμε αυτό το θέμα. Από τη μία πλευρά είμαστε ευχαριστημένοι που υπάρχει λόγω της πυκνής προσφοράς ε, και περισσότερη επιλογή ε, και οι καταναλωτές έχουν περισσότερο χρόνο να ψωνίσουν ε, λόγω του διευρυμένου ωραρίου ε, και εμείς το ξέρουμε αυτό πάρα πολύ καλά αυτό το πλεονέκτημα μπορούμε να ψωνίσουμε στις 8, 9, 10 το βράδυ ε, Βεβαίω αυτό το παρατεταμένο ωράριο καταβροχθίζει Πολύ ενέργεια και δημιουργεί και πάρα πολλά απορρίμματα. Εάν δηλαδή πρέπει να είναι ανοιχτά τα καταστήματα, ιδίω τροφίμων μέχρι τις 9-10 το βράδυ, ε, στο τέλος ε, πετιούνται ως απορρίμματα τα τρόφιμα τα οποία δεν μπορούν να πουληθούν την επόμενη μέρα, φρέσκα. Λοιπόν, αυτή η, ο, τρύπο, ο τύπος της ε, κατανάλωσης, ε, την οποία αποκαλούμε ας πούμε αηφόρο, ήταν μια καλή ιδέα. Έχει όμως ε, και την αντίστροφη πλευρά, την άλλη πλευρά του νομίσματος και πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τα αρνητικά. Λέμε λοιπόν τώρα ότι θέλουμε να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα δράσης ε, για αυτήν την κατανάλωση, ε, αλλά όταν σκεφτόμαστε το θέμα της αηφορίας, της διάρκειας, ε, της αένταης κατανάλωσης αν θέλετε, πρέπει να σκεφτούμε και τα αρνητικά, τις αρνητικές επιπτώσεις. Άρα λοιπόν, πούμε να επιτύχουμε τους στρατηγικούς στόχους του 2020, έχουμε πάρα πολύ δουλειά μπροστά μας. Επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί θα, πρέπει οι χώρες προμηθευτές να είναι στην πρώτη γραμμή. Ωραία θα ήταν να ήταν στην πρώτη γραμμή των στόχων μας, αλλά να μην ξεχνάμε και τους πελάτες. Δεν είναι μόνο η προσφορά, αλλά είναι και η ζήτηση ε, που πρέπει να προσέξουμε. Ένα άλλο σημείο το οποίο πιστεύω δεν έχει καλυφθεί επαρκώς είναι το άνοιγμα στις επιχειρήσεις και στους καταναλωτές. Αναφέρατε το θέμα της ε, έδρας ε, αλλά εδώ έχουμε τρεις πτυχές που πρέπει να προσέξουμε. Ε, της χωροταξίας ε, πρέπει να προσέξουμε ώστε να μην απονεκρωθούν ε, οι εσωτερικές περιοχές των πόλεων, τα κέντρα δηλαδή των πόλεων και να χτίζονται καινούργια καταστήματα και πολυκαταστήματα μόνο στην περιφέρεια. Πρέπει λοιπόν και το χωροταξικό αστικό ε, σχέδιο, το προγραμματισμός να προσεχτεί επαρκώς. Επίσης το ηλεκτρονικό εμπόριο, το e-commerce, ε, μειονεκτεί σημαντικότατα στην, στην Ήπεθρο. Είναι πολύ δύσκολο ε, σε αγροτικές περιφέρειες πιο ηλικιωμένοι άνθρωποι και δι γυναίκες να εκμεταλλευτούν τα πλανεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πώς θα λύσουμε το θέμα της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ήπεθρο και στις αγροτικές περιοχές. Ε, πολλοί υπεραμείνονται του τοπικού ε, μπακάλικου, τον μπακαλικάκι α πούμε του χωριού. Μήπως πρέπει να υποστηρίξουμε αυτό και να επιλέξουμε εναλλακτικές λύσεις ε, και να προσέξουμε να μην απονεκρωθούν, να μην ερημωθούν αυτές οι περιοχές. Πρέπει λοιπόν να ενισχυθούν όλες οι μορφές κατανάλωσης και να είναι ευέλικτοι οι κανόνες που θα προτείνει η Κομισιόν. Τώρα, όσον αφορά τις ευέλικτες μορφές εργασίας, πολλά μπορούν να γίνουν. Και πάλι όμως υπάρχει η αντίστροφη πλευρά του νομίσματος. Υπάρχει η κακή κατάρτιση, η ανεπαρκής κατάρτιση, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι που περνάνε από ένα πρόγραμμα κατάρτισης να μην εκπαιδεύονται καλά και σωστά. Άρα λοιπόν είναι δύσκολο να πείσουμε τους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις να επενδύσουν, να ξοδέψουν περισσότερα για την κατάρτιση του προσωπικού αν, και, αν τα προγράμματα δεν είναι ικανοποιητικά. Ευχαριστώ κυρία Ρίλε, λέει πρόεδρος, ο επόμενος ε, μιλητής είναι ο πρόεδρος, ο κύριος Χάρμπορ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είμαι σκιώδης εισηγητής για την ομάδα μου στην έκθεση της Άννας Μαρία. Μαρίας. Και ε, πιστεύω ότι αυτό το οποίο έχει κάνει μέχρι τώρα δικαιολογεί απόλυτα την απόφαση ε, για μια έκθεση πρωτοβουλίας. Είναι σημαντικό να προχωρήσουμε αυτά τα θέματα και μέσω της ακρόασης και με την εργασία που έχει κάνει αναπτύσσεται ο διάλογος με ένα πολύ σημαντικό τομέα. Uh, ένα πάρα πολύ, μια πάρα πολύ ανταγωνιστική αγορά λιανικού εμπορίου όπου η αλυσίδα προμηθειών είναι θεμελιώδης, είναι θεμελιώδης για να ενισχύσει μία από τη επιτυχημένη, ανταγωνιστική και διαφοροποιημένη λιανική αγορά. Έχει λοιπόν πολλές πτυχές αυτό το ζήτημα και απαιτεί θάρρος από την εισηγήτρια να να μελετήσει όλα αυτά τα ζητήματα και το, το θάρρος αυτό το έχει δείξει η εισηγήτρια. Όσον αφορά τη δική μου συμβολή και την ισορροπία της ε, έκθεσης, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να μην υποτιμήσουμε το γεγονός ότι έχουν γίνει τεράστιες επενδύσεις στο λιανεμπόριο σε όλη την Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την ε, παράδοση ε, και τη διακίνηση αγαθών με νέες μορφές νέα προϊόντα, νέοι τρόποι διανομής, παράδοσης κλπ. Και εάν θέλουμε να παρέμβουμε, πρέπει να παρέμβουμε ελαφρά, προσεκτικά. Να μην υπονομεύσουμε τη δυναμικότητα και την ε, ανάπτυξη αυτού του τομέα υπάρχουν διαδικασίες στο λιανικό εμπόριο οι οποίες είναι πρωτοπόρες ε, στο διεθνές επίπεδο και δεν πρέπει να τις υπονομεύσουμε ή να τις περιορίσουμε. Υπάρχουν εξαιρετικά επιτυχημένες διεθνείς εταιρείες λιανικού εμπορίου που εδρεύουν στην Ευρώπη αλλά δραστηριοποιούνται σημαντικότητα στην Κίνα, στις Ηνωμένε Πολιτείες και αλλού. Είναι διεθνείς παίκτες. Τώρα, οι, το, οι δυνατότητες αυτές ε, μπορούν να προσφερθούν εφόσον έχουν μια εξαιρετική διαχείριση της αλυσίδας προμηθειών. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να τονίσουμε σε αυτή την έκθεση ότι εάν θέλει κάποιος να έχει μια εξαιρετικά επιτυχημένη επιχείρηση λιανικού εμπορίου, δεν είναι μόνο, δεν πρέπει μόνο να είναι επιτυχημένος στην πλευρά της παράδοσης των προϊόντων, των παραγγελιών, αλλά και στην πλευρά της προμήθειας. Να έχει δηλαδή ένα πάρα πολύ σωστό δίκτυο προμήθειας των προϊόντων, τα οποία θέλει να πουλήσει. Και η συγγήτρια λέει πάρα πολύ σωστά ότι υπάρχουν θαυμάσιες ευκαιρίες δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και κατάρτισης εκπαίδευσης σε όλη την αλυσίδα του λιανικού εμπορίου. Η κυρία Κοράτσο Μπίλτ έχει ακριβώς τονίσει αυτή τη σημασία της αλυσίδας προμηθειών. Τώρα, υπάρχουν ορισμένες ε, πτυχές της έκθεσης που μπορούμε να προσθέσουμε αξία το ανταγωνιστικό λιανεμπόριο ενισχύεται με την ε, εφαρμογή νέων τεχνολογιών αλλά και πράσινων διαδικασιών. Πρέπει να ενισχύουμε λοιπόν και τις πράσινες διαδικασίες. Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι ορισμένες ε, αλυσίδες, ε, ορισμένοι κόμβοι του λιανικού εμπορίου έχουν απομακρυνθεί από τη διαμόρφωση της πολιτικής εδώ στις Βρυξέλλες. Αυτό που θέλουμε είναι η πολιτική που μελετάμε εδώ να είναι κοντά στο λιανικό εμπόριο έτσι ώστε μαζί να μπορούμε να βρούμε νέες μεθόδους και νέους τρόπους εργασίας. Ήδη έχουμε κάνει ενδιαφέρουσες συζητήσεις με, τους, ε, με, με, τις, με τα μεγάλα πολυκαταστήματα λιανικού εμπορίου DIY, δηλαδή αυτά που ε, φτιάχνεις μόνος σου τα κατασκευαστικά πολυκαταστήματα και μπορούμε μπορούμε συνεργαζόμενοι με τους προμηθευτές, με τα πολυκαταστήματα αυτά που πουλάνε οικοδομικά, υλικά κλπ, να βελτιώσουμε την, ε, τον κατασκευαστικό τομέα των σπιτιών. Παραδείγματο χάρη να ενισχύσουμε τα πράσινα υλικά, τις πράσινες διαδικασίες και να βελτιώσουμε τον ε, οικιστικό τομέα. Υπάρχουν όμως και άλλες ε, περιοχές, άλλοι τομείς όπου μπορούμε να προωθήσουμε την τεχνολογία. Ξέρουμε ότι και σε άλλους ε, τομείς όπως την ε, ταυτοποίηση ε, προϊόντων ραδιοσυχνοτήτων μπορούμε να προσφέρουμε στους καταναλωτές πληροφορίες και δυνατότητα ανείχνευσης των προϊόντων που αγοράζουν. Ανιχνευσιμότητα και ποικιλία Ξέρουμε βεβαίως ότι η προσωπική συμπερι... η καταναλωτική συμπεριφορά παρακολουθείται. Δηλαδή υπάρχουν ε, συστήματα τα οποία παρακολουθούν αυτά τα οποία αγοράζουν οι ιδιώτες και πότε και ποια προϊόντα. Ε, πρέπει λοιπόν και αυτό να το συμπεριλάβουμε στην εξέταση της ενιαίας αγοράς ε, από μια ολιστική άποψη, δηλαδή όλες τις ψυχές να τις συμπεριλάβουμε. Εξετάζουμε το ρόλο των λιανών πολιτών, των προμηθευτών, ε, για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Ε, ταυτόχρονα θέλουμε να βελτιωθεί η πράσινη πτυχή, να είναι ευέλικτη η αγορά και να έχει μεγάλη διείσδυση. Θα υποβάλω λοιπόν ε, σχετικές τροπολογίες. Και τέλος, ε, η πράξη αυτή της ενιαίας αγοράς ε, Έχουμε ήδη υποβάλει μερικές τροπολογίες οι οποίες συνδέουν την πρόταση της κυρίας Μπίλτ με την πράξη της ενιαίας αγοράς και πιστεύουμε ότι στην τελική πρόταση για την πράξη της ενιαίας αγοράς θα ληφθούν υπόψη αυτές οι τροπολογίες που έχουμε υποβάλει και θα συζητηθούν αύριο το απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Ο Κυριάκος Τενταφυλίδης είναι επόμενος. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ την εισηγήτρια για τη σε εργασία που έχει κάνει να τη διαβεβαιώσω ότι θα συνεργαστούμε μαζί της στις επόμενες συναντήσεις με τους ε, Shadow Rapporteurs. Ωστόσο, σαν ομάδα της αριστεράς, εμείς τασόμαστε κριτικά απέναντι στα βασικά σημεία της έκθεσης, γιατί κατά την άποψή μας δεν έχει μια ισοζυγισμένη προσέγγιση στην οποία κεντρικό ρόλο θα έχουν και οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προτείνει για παράδειγμα λύσεις περιττέρω ανοίγματο των αγορών και συγκεντρωποίηση τους στα μεγάλα αστικά κέντρα, χτυπώντα κατά την άποψή μας τον πυρήνα της λιανικής αγοράς, δηλαδή τον μεμονωμένο παραγωγό. Ταυτόχρονα είναι κεντρική σημασία στο ζήτημα της απόκληση των τιμών και η αντιμετώπιση του, σημείο στο οποίο θα επανέλθουμε αργότερα με προτάσεις τροπολογιών. Αναλυτικότερα Όσο αφορά το κεφάλαιο καθιστώντας την πρόσβαση στην αγορά πιο προσιτή για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές και την παράγραφο 14 γίνεται νήξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε σχέση με τις τοπικές αγορές και τα τοπικά καταστήματα τα οποία μειώνονται προς όφελος των μεγάλων εμπορικών κέντρων. Εδώ παρουσιάζεται μια αδυναμία να προταθούν ουσιαστικά μέτρα για στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είμαστε της άποψης ότι η Κομισιόν θα πρέπει να ενισχύσει τις προσπάθειες των κρατών μελών για προώθηση αντισταθμιστικών μέτρων στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προσφέροντας έτσι όχι μόνο θέσεις εργασίας, αλλά και καλύτερη πρόσβαση των καταναλωτών σε ποιοτικά και οικονομικά προσιτά προϊόντα. Επίσης θα ήθελα να σταθώ στο σημείο σχετικά με τη δύναμη των επιχειρήσεων στην αγορά του λιανεμπορίου. Ορθά η εισηγήτρια σημειώνει τους κινδύνους δεσπόζουσας θέσης από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και προς τούτο θα πρέπει ακριβώς τα μέτρα και οι προτάσεις που κατατίθενται να μην ενισχύουν αυτούς τους κινδύνους. Συμπληρωματικά αξίζει να πούμε ότι ακριβώς η ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης από μεγάλες επιχειρήσεις είναι ένας από τους παράγοντες που συμβάλλουν στην απόκληση τιμών που παρουσιάζεται στη λιανική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, κυρία Πρόεδρε, για τους μισθωτούς, η βασική πολιτική κατεύθυνση που θα πρέπει να μας χαρακτηρίζει είναι ο σεβασμός των συλλογικών συμβάσεων και των δικαιωμάτων τους και η στόχευση ενός αξιοπρεπούς βιωτικού επίπεδου και κατ' επέκταση ενός αξιοπρεπούς μισθού. Ευχαριστώ πάρα πολύ και όπως είπα θα επανέλθουμε με τροπολογίες και θα συνεργαστούμε στις συναντήσεις που θα γίνουν με τους ε, shadow rapporteurs. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ας δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κ. Μπέρκοβε. Ε, <clears throat> Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω ευχαριστώντας την εισηγήτρια. Ήταν έξοχη η συνεργασία μας, επί μήνες. Ευχαριστώ και τους Σκιώδης. Καλωσορίζουμε την έκθεση που υποβάλλεται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως γνωρίζετε, προσπάθησε να ακολουθήσει στις δικές της εκθέσεις της ολιστική προσέγγιση, υπογράμμισε κάποια ζητήματα. Είναι πολύ ενθαρρυντικό που βλέπουμε ότι η Επιτροπή σας, η συγήτρια και η σκιώδης, συμφωνούν ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί ολιστική προσέγγιση και πολλά βασικά θέματα υπογραμμίστηκαν. Να πω επίσης, σχετικά με αυτό, ότι η έννοια ενό ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για τον τομέα του λιανικού εμπορίου είναι κάτι ευπρόσδεκτο από εμά. Αναφέρθηκαν διάφορα στοιχεία και από την εισηγήτρια και από τους σκιώδεις. Διάφορα θέματα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στη στρατηγική αυτή. Όσον αφορά την καινοτομία, πράγματι φρονούμε ότι αυτός ο τομέας όχι είναι μόνο σημαντικός για την απασχόληση, αλλά δράει και σαν κόμβος για την εσωτερική αγορά, λόγω της αλυσίδας ε, τροφοδοσίας των προϊόντων. Ε, προσπαθούμε λοιπόν να έχουμε εύρυθμη εσωτερική αγορά. Ευπρόσδεκτο κάτι που είναι γνωστό στην Επιτροπή και την ενδιαφέρει. Δηλαδή το ηλεκτρονικό εμπόριο θα πρέπει να θεωρηθεί ως βασικό συμπλήρωμα των δραστηριοτήτων του τομέα του λιανικού εμπορίου. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό στα δραστηριότητα, θα γνωρίζετε οι περισσότεροι ότι πολλοί, μερικοί μάλλον, πολύ ανταγωνιστικοί για πολιτέ ε, εκπροσώποι του ελληνικού εμπορίου ε, κινούνται μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να ληφθεί υπόψη. Προσπαθώ να είμαι όσο θετικό γίνεται. Διότι μετά πρέπει να απαντήσω στο ένα ερώτημα που έθεσε η πρόεδρό σα, το οποίο σύθιστε δεν μπορώ να απαντήσω. Ε, τι εμπεριέχεται στην πράξη για την ενιαία αγορά. Άκουσα προσεκτικά, αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω, και θα συναντηθώ με τον Επίτροπό μου ε, το απόγευμα και θα διαβιβάσω το ενδιαφέρον ε, της Επιτροπής σας για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Τέλος, κάτι εξίσου σημαντικό, είναι ευαίσθητο το ζήτημα των ε, συμβασικών σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων και σχετικές πρακτικές που ακολουθούνται. Ε, όπως γνωρίζει το Κοινοβούλιο, ήταν επίμαχο θέμα, κυρίως στα πλαίσια της τροφικής αλυσίδας, ε, υπάρχουν πολλές εκθέσεις σχετικές. Πιέστηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιδράσει. Διεξάγεται συζήτηση τώρα, όπως εξήγησαν εξηγείται και η κυρία Κοράτσα Μπίλτ με τους εμπλεκομένους φορείς στην ομάδα υψηλού πιπέδου για τα τρόφιμα. Είναι ένας φορέας που εξετάζει το θέμα αυτό και οι εμπλεκόμενοι καταβάλουν προσπάθειες για να συνομιλήσουν, να συνεννοηθούν να συμφωνήσουν επί βασικών αρχών. Για να το πετύχουν αυτό, και αυτό είναι σημαντικό για το χρονισμό, για να το πετύχουν αυτό ελπίζουμε να καταλήξουν κάπου προς το τέλος του έτους. Και όπως είπαν και αρκετά μέλη, εμείς δεν θέλουμε να προδικάσουμε τα αποτελέσματα των εν λόγω συζητήσεων, προτείνοντας κάποια πρωτοβουλία σε πρώιμο στάδιο. Τι προτείνουμε λοιπόν, μια ανακοίνωση για το φθινόπωρο. Και τι θα κάνουμε με αυτό δηλαδή. Θα προσπαθήσουμε να ανανεώσουμε την προβληματική σε οριζόντιο επίπεδο, διότι αυτό είναι κάτι που ετέθη για την τροφική αλυσίδα. Ε, είναι ευρύτερο όμω θέμα, όπως γνωρίζετε, δεν αφορά μόνο το λιανικό εμπόριο, είναι ένα θέμα μικρομεσών επιχειρήσεων. Και θέλουμε να εκθέσουμε ξεκάθαρα το θέμα αυτό στην επικείμενη ανακοίνωσή μας και να κάνουμε κάτι που δυστυχώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έκανε ακόμα και θα έπρεπε να το κάνει. Ήτι να χαρτογραφήσουμε το τι εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση του προβλήματο. Είτε στα πλαίσια περί ανταγωνισμού, αθεμή του ανταγωνισμού και αυτό που είπε η κυρία Κοράτσα Μπίλτ και συστήματα αυτοεπιβολή, αυτοσυμμόρφωσης αν θέλετε που σε κάποιου τομεί, από ό,τι ακούμε τουλάχιστον, είναι συστήματα που μπορούν να λειτουργήσουν αρκετά αποτελεσματικά επουδενή δεν διατηνόμεθα ότι δεν είναι σημαντικό το ζήτημα. Συμφωνούμε όμως με το γενικό πνεύμα της εκθέσεως. Δηλαδή, θα πρέπει να το εξετάσουμε προσεκτικότατα πριν αποφασίσουμε τι είδους ευρωπαϊκή δράση απαιτείται, αν απαιτείται τέτοια. Και να ενθαρρύνουμε πραγματικά τα εμπλεκόμενα μέρη να καταλήξουν σε αποτελεσματικότερες και πιο θεμητές επαγγελματικές ε, πρακτικές. Επικερδές για όλους, βιωσιμότητα, επιλογή καταναλωτών, καινοτομία, επενδύσεις. Σε αυτό το στάδιο βρισκόμαστε όσον αφορά αυτή την πρωτοβουλία και με τα χαράς να απαντήσω σε περαιτέρω ερωτήσεις αν αυτές υπάρχουν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Κορότσα τώρα. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να περάσω κάποια πολύ σημαντικά θέματα που ανέφεραν οι συνάδελφοι. Να ευχαριστήσω και πάλι την Κομισιόν για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε. Χαίρομαι που προχωρήσαμε τόσο πολύ. Ε, φίλος μου Παντσέρη, φίλε μου Παντσέρη, είναι σημαντικό να σεβαστούμε το θέμα της επικουρικότητας και προσπάθησα να επικεντρωθώ σε αυτό, σε την ε, έκθεση για το πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά σε επίπεδο κοινότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το αν μπούμε στη σχέση των ε, συλλογικών συμβάσεων ε, και των σχέσεων εργοδότη και εργαζόμενου, δεν ξέρω αν πρέπει να το χειριστούμε αυτό σε, σε επίπεδο ένωσης. Αλλά είναι καλό να ενθαρρύνουμε τον κλάδο των εργοδοτών να ε, βελτιώσουν την κοινωνική και εταιρική ευθύνη. Επίσης, το θέμα του περιβάλλοντος. Εγώ ήδη ε, η ίδια εκπλάγει θετικά με το πόσες θετικές δράσεις έχουν ε, ήδη ληφθεί, πόσες πρωτοβουλίες, πόσα φόρουμ για την βιώσιμη ανεφόρο κατανάλωση και ο διάλογος πολλές φορές ξεκινάει από τον ίδιο τον κλάδο των εργοδοτών. Πρέπει να υπάρξει ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών και βλέπω ότι ήδη γι' αυτό γίνεται. Και να το υποστηρίξουμε. Το εταιρικό μοντέλο το έχουμε δουλέψει στη διαβούλευση με τη, με Eurocop, ε, ήταν στο πάνελ μαζί μας και ξέρουμε την προσθεμινή του θέματος. Δεν ξέρω αν η τροπολογία εδώ α, ταιριάζει εδώ πέρα, αλλά είμαστε ανοιχτοί σε αυτό. Τώρα για το Μάρτεν Λόκεγκάρτ, το συνάδελφο από την Άλντε. Από το Άλντε. Συμφωνούμε ασφαλώς ότι η επιβολή είναι προτεραιότητα. Πριν ζητήσουμε νέα νομοθεσία πρέπει να δούμε τις επιλογέ που έχουμε ήδη στη διάθεσή μα και θα πρέπει η Κομισιόν να μα το ξεκαθαρίσει αυτό. Κυρία Ρούλε, ευχαριστώ πολύ. Να πω ότι είχα βάλει το θέμα της πράσινη σήμανση, οικολογική σήμανση, αλλά το, τελικά το αφαιρέσαμε για λόγω έλλειψη χώρου. Αλλά θα ήθελα να δω την τροπολογία της κυρίας Ρούλε. Η αεφόρου κατανάλωση είναι στο κέντρο τη. Ε, ατζέντα και νομίζω ότι αυτό ελπίζω ότι είναι αντανακλάται στην έκθεση. Είναι κεφαλαίου σημασία. Οι επιχειρηματίε έχουν μεγάλη ευθύνη στο να προωθήσουν ε, και, ε, καινοτόμα προϊόντα τα οποία είναι πιο αναργιακά αποδοτικά και δημιουργούν λιγότερα απόβλητα. Στο σχέδιο δράσης τώρα θα, είναι, θα προτείνουμε εμείς στην Κομισιόν να περιλάβει ένα σημείο για την φόρο κατανάλωση λοιπόν. Όταν λέτε ότι δεν υποστηρίζετε το γεγονός ότι η, η πλευρά του εφοδιασμού είναι, ε, θα είναι πρωτοφόρη σε αυτό το θέμα, εγώ κατά τη γνώμη μου έχουν κεντρικό ρόλο στο να ε, στη μάχη ενάντια στη, στο διαβήτη και γενικά υπέρ του, της σωστής διατροφής. Τώρα για τον συνάδελφο από, την από τον ΚΟΕ. Ε, αν δεν ξέρω αν να διευκρινίσετε, εκεί που είπατε ότι η έκθεση οδηγεί στην περιττέρω ενίσχυση των αστικών περιοχών. Δεν ήταν αυτό που ήθελα εγώ να πω. Θεωρώ ότι κάτι πρέπει να γίνει για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ που το αναφέρατε το θέμα της το θέμα των τοπικών αγορών, των τοπικών μικρών μαγαζιών σε αντίθεση με τα μεγάλα εμπορικά κέντρα ή τα one-stop shop. Ζητώ από την Κομισιόν να το εξετάσει το θέμα πρέπει να υπάρχει ο απαραίτητο διάλογο μεταξύ των ε, δημιουργών εμπορικών κέντρων και των ε, ε, ιδιοκτητών των, των Υπάρχει ένας διάλογος και στη Σουηδία γι' αυτό. Δεν ξέρω αν τα αντισταθμιστικά μέτρα είναι ο καλύτερος τρόπος να ενισχύσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά μπορούμε να το εξετάσουμε. Μάλκο, με ευχαριστώ για την υποστήριξή σου και καλά σου λόγια. Θα συμφωνούσα ότι πρέπει να βάλουμε την καινοτομία στο επίκεντρο α, της έκθεσης και ε, να το διευρύνουμε το θέμα πέρα από τα θέματα ανταγωνιστικότητας. Το θέμα των α, ε, υψηλών δεξιοτήτων δεν είναι μόνο α, ε, απασχόληση για άτομα με χαμηλές δεξιότητες, αλλά και με υψηλές δεξιότητες. Καλό θα ήταν να ενθαρρύνουμε τους ε, λιανέμπορους να, να βοηθούν στο θέμα της επιμόρφωσης, της ανάπτυξης των δεξιοτήτων και θα θέλω να ακούσω τις τροπολογίες. Τώρα, το κατά πόσο το λιανικό εμπόριο είναι προτεραιότητα για την Κομισιόν. Να πω ότι με την ε, υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού και χαίρομαι που υπάρχει και η πλήρης υποστήριξη του κύριου Χάρμπορ. Έχουμε ζητήσει να ληφθεί υπόψη στις προτεραιότητες στο νόμο για την εννέα αγορά. Μέχρι στιγμή ήταν πολύ θετική ανταπόκριση από την Κομισιόν και να σας ευχαριστήσω για αυτή την υποστήριξη. Είμαι ανοιχτή σε περαιτέρω ερωτήσεις και θα ήθελα να συναντήσω και τους σκιώδους συζητητές. Τέλος να πω ότι ζούμε σε εποχή μεγαλύτερου προστατευτισμού. Και η Ευρώπη δεν ανταγωνίζεται στο, στην παγκόσμια αγορά. Νομίζω ότι ε, έχουμε μεγάλη ευθύνη ε, με, την έκθεση αυτή να πούμε ότι και η Ευρώπη πρέπει να έχει φιλοδεξία να είναι πρωταθλήτρια στην ε, παγκόσμια αγορά και να, παρασ... και να, να παράσχει περισσότερες δουλειές στο κλάδο του λιανεμπορίου. Ευχαριστώ. Η κατάσταση τροπολογιών προθεσμία είναι 19 Απριλίου το 12 η ώρα και η ψηφοφορία 25 Μαΐου. 19 Απριλίου, 25 Μαΐου. Και προχωρούμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξη και καλό τον πρόεδρο Α, λύεται η συνεδρίαση, λέει η προεδρεύουσα. Ε, ακόμα καλύτερα, ακόμα καλύτερα. Και παρακαλώ να επανέλθετε το απόγευμα. Θα, συζητήσουμε την έκθεση Παντσέρη. Α, έχουμε μία ακρόαση. Για τα αγροτικά μηχανήματα. Ακρόαση το απόγευμα για τα αγροτικά μηχανήματα. Παρακαλώ, ελάτε.